διεθνής συνεδρίασης διατίθενται εάν τα θέλετε δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υιοθετήθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης ε,